Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεθνής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τότε τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Σας ευχαριστώ. Μία ανακοίνωση μόνο.